καταστήσω γνωστό ότι στις 7 Απριλίου έλαβα επιστολή του κύριου Φάρετς, συμπροέδρου της Ομάδας Ευρώπη και Δημοκρατίας. Καλείται το σημείο 6 του κανονισμού, το άρθρο 6 μάλλον, και ε, διαμαρτύρεται για τον τρόπο ε, με τον οποίο χειριζόμαστε στην Ευρώπη τις ε, ε, βουλευτικές ασυλίες. Διαβίβασα το αίτημά του στην Νομική Επιτροπή. Έρχομαι τώρα στην ημερήσια διάταξη να σας παρουσιάσω. Την έχετε στα χέρια σας και να δούμε την κάθε μέρα ξεχωριστά. Διαδικαστικό.